Ε, η μερίστη διάταξη που είχατε λάβει αφορούσε την συζήτηση για την τελευταία ΚΟΖΑΚ υπό τη Βελγική Προεδρία. Αλλά η συνεδρία των συντονιστών θεώρησε σκόπιμο να την αναβάλει αυτή τη συζήτηση για άλλη ημερομηνία, γιατί θα θέλαμε να είναι παρόν όχι μόνο ο συμπρόεδρος, εγώ δηλαδή υποφαινόμενος, μαζί με τον κύριο Μαρτίνες της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ε, ο Μαρτίνες που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αφαιρέθηκε λοιπόν αυτό το σημείο από την ημερήσια διάταξη και ανεβλήθηκε για μια επόμενη συνεδρίαση. Το υπόλοιπο σχέδιο της ημερήσιας διάταξης το λάβατε στις 28 Οκτωβρίου με τις διορθώσεις που σας ανέφερα. Νομίζω πως ε, θα μπορέσετε κι εσείς να το εγκρίνετε. Ε, λοιπόν, ανακοινώσει του Προέδρου. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια επιστολή, το ανέφερα και στους συντονιστέ, μια επιστολή που ε, μας έστειλε ε, η Προεδρία μέσω του κυρίου Σαστέλ στον Πρόεδρο Μπούζικ, όπου εκφράζονται επιφυλάξει γενικού περιεχομένου σε σχέση με την συμφωνία πλαίσιο που συνήφθη μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ε, κατ' ουσίαν ο Προεδρεύων Σαστέλ δηλώνει ότι η θεσμική ισορροπία θα πρέπει να ε, γίνει αυστηρά σεβαστή και ότι αν ε, παραβιαστεί το Συμβούλιο δεν θα διστάσει να προστρέξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι μια ανακοίνωση προληπτικού χαρακτήρα, δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο και οι συντονιστέ θεωρούν ότι θα πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν, να δούμε τι θα γίνει και την κατάλληλη στιγμή να ενεργήσουμε με την απαραίτητη αποφασιστικότητα. Να θυμίσω ότι στις 21 Οκτωβρίου ε, που μας πέρασε υπήρξε μια συνάντηση μιας αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου Δηλαδή, εγώ, η Αντιπρόεδρος Γκουρμάη και η κυρία Τέιν και Λεγκρίπ είχαμε μία επαφή λοιπόν με μια ομάδα βουλευτών από την Νότια Αφρική που επισκέφθηκαν εδώ το Κοινοβούλιο και που θέλησαν να συναντήσουν την Επιτροπή μας. Δεν υπήρχε συνεδρία της Επιτροπής και γι' αυτό και ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήταν παρόντες, θέλησαν μάλλον να συμμετάσχουν σε αυτήν την συνάντηση με μια πολυάριθμη αντιπροσωπεία της Νότιας Αφρικής. Ήταν 15-16 βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων της χώρας τους το Κοινοβουλίου της χώρας τους και μας ρώτησαν πληροφορίες για το πώς ελέγχουμε το εκτελεστικό, πώς ε, μεταρρυθμίζονται οι συνθήκες και ούτω καθεξής, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το εξή. Στην Νότια Αφρική υπάρχει ένα σύνταγμα που ισχύει από το 1996 και που προβλέπει ότι ετησίως μπορεί να υποβληθεί σε μεταρρύθμιση. Και ε, είναι μια ειδική επιτροπή Υπάρχει μια επιτροπή ειδική για τη μεταρρύθμιση του συντάγματος. Οι βουλευτές λοιπόν που ήρθαν εδώ ήταν ε, αυτοί που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη επιτροπή. Ήθελαν να δουν λοιπόν τι μπορούμε εμεί να τους προτείνουμε για μια ενδεχόμενη μεταρρύθμιση του συντάγματός του. Είναι προφανέ ότι σε μια συνάντηση μια ώρα δεν είναι δυνατόν να του πούμε και πολλά πράγματα. Ανταλλάξαμε κάποιε πληροφορίε, ε, αγγίξαμε και το θέμα τη ε, νομική. Ε, ανεξαρτησίας του νομικού σώματος, ε, του δικαστικού σώματος, συγγνώμη, αλλά ήταν απλώς ε, μια συζήτηση ενδιαφέρουσα βέβαια, αλλά γενική. Η ομάδα των συντονιστών πριν από λίγο αποφάσισε για να δώσει μια κατεύθυνση σε αυτά τα αιτήματα ε, που μας έρχονται από βουλευτές άλλων χωρών, δηλαδή να είμαστε ανοιχτοί, να υποδείξουμε ως ημέρα συνάντησης με τέτοιες αντιπροσωπείες μια μέρα που συνεδριάζει και η Επιτροπή μας και αν αυτό δεν είναι δυνατόν να αναζητούμε την να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση με παρουσία των μελών της Επιτροπής μας. Να μην είναι μόνο ένας άνθρωπος δηλαδή που θα τους δεχτεί, να είμαστε τουλάχιστον πέντε όταν έχουμε τέτοιες επισκέψεις. Αυθορμήτως πώς λοιπόν αυτή τη φορά στην ουσία θέσαμε σε εφαρμογή αυτά που αποφάσισαν με κατόπιν εορτής οι συντονιστές. Να σας πω επίσης ότι στις τελευταίες συνεδρίες των συντονιστών, δηλαδή την προηγούμενη, όχι τη σημερινή, την προηγούμενη φτάσαμε σε μια συμβαστική συμφωνία σε σχέση με την έκθεση του συναδέλφου Ντάφ για την εκλογική διαδικασία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα και τα πιο περίπλοκα ζητήματα που εξετάζουμε. Ε, συγκεκριμένο αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας είναι μια νέα εκδοχή της έκθεσης του συναδέλφου Νταφ που αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στα αγγλικά και σε αυτή τη γλώσσα διανεμήθησε σε όλους αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατή η μετάφραση στις άλλες γλώσσες ακόμη. Προβλέπεται λοιπόν η συζήτηση για την επόμενη συνεδρίαση στις 29 και 30 Νοεμβρίου. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο έγγραφο του συναδέλφου Νταφ που σχετίζεται με τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Και αυτό το έγγραφο το έχει ετοιμάσει ο κύριος Νταφ. Πάλι μόνο στα αγγλικά το έχουμε. Δυστυχώς η μετάφραση δεν έχει γίνει ακόμη και θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας 29 και 30 ε, Νοεμβρίου 2010. Τώρα, για την πρωτοβουλία των πολιτών θα μιλήσουμε αύριο και άρα πρέπει εγώ να σας πω δύο λόγια για την ερμηνεία που πρέπει να δώσουμε στο άρθρο 51 του κανονισμού μας. Το ζήτημα δεν είναι και τόσο απλό όσο φαίνεται καταρχήν. Και γι' αυτό σήμερα σας παρουσιάζω ένα έγγραφο εργασία που σας έχει ήδη διανεμηθεί. Ελπίζω να το έχετε διαβάσει και παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα ερμηνείας του κανονισμού μας. Για την ώρα θα πρέπει να λάβετε υπόψη πως αυτή τη δικασία του άρθρου 51 έχει εφαρμοστεί λίγες φορές. και απαιτείται ε, μετά από την πρώτη ανάγνωση ε, των νομοθετικών ε, κειμένων. Άρα λοιπόν οι συνάδελφοι πρόεδροι των Επιτροπών μας ζήτησαν να γνωμοδοτήσουμε. Ζητήθηκε και από τον πρόεδρο Λένε, από την Επιτροπή δηλαδή Περιβάλλοντος και από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να γνωμοδοτήσουν. Και εκείνοι υπέδειξαν κάποιες δυσκολίες ερμηνείας. Στην ουσία να σας πω περί τίνος πρόκειται. Ο συνάδελφος Λένεν, να σας πω καταρχήν το ιστορικό. Ήδη γνωρίζετε πως είναι δύσκολα τα πράγματα, λοιπόν γνωρίζετε. Η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές στη νομοθετική εργασία διέπεται από τα άρθρα 49, 50 και 51 του κανονισμού. Το άρθρο 49 προβλέπει την φυσιολογική κατάσταση όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή που ορίζεται ω αρμόδια επί τη ουσία, αλλά μπορεί να υπάρχουν μια και περισσότερε επιτροπέ που δίνουν μια γνωμοδότηση. Το νόημα αυτή τη γνωμοδότηση και ο ρόλο των επιτροπών αυτών ρυθμίζεται από το 49. Λοιπόν, το 51 τώρα περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία κάποια συγκεκριμένη έκθεση εμπίπτει στις αρμοδιότητες όχι μόνο μιας επιτροπής, αλλά περισσότερων. Και αυτή η διπλή αρμοδιότητα μπορεί να αφορά ολόκληρο το κείμενο Άρα είναι και δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων μια επιτροπή και των αρμοδιοτήτων μια άλλη, αλλά μπορεί επίση να αφορά μεμονωμένα τμήματα κάποια έκθεση, όπου α πούμε μπορεί κάποιο τμήμα να εμπίπτει απόλυτα στι αρμοδιότητε τη επιτροπή που έχει οριστεί ω αρμόδιο από τη ουσία, αλλά και κάποια άλλα τμήματα σε άλλε αρμοδιότητε άλλων επιτροπών. Και το 51 ρυθμίζει τα πράγματα λέγοντα ότι τα κομμάτια αυτά που αφορούν ε, αρμοδιότητες άλλων επιτροπών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών που δεν ψηφίζονται στην Επιτροπή αλλά μπορούν να υποβληθούν άμεσα στην Ολομέλεια και προβλέπει επίσης ότι στην ε, δεχόμενη περίπτωση μιας ε, συνδιαλλαγής οι εισηγητές της συνδεδεμένης αυτής της μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες. Το 51 λοιπόν μιλά για κάτι ακόμα. Λέει λοιπόν ότι εφόσον ε, πληρούνται οι όροι που εκτίθενται στο άρθρο 49 παράγραφος 1, πράγμα το οποίο δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί αυτό ε, αφορά τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιτροπών, πράγμα το οποίο υπονοεί τις περιπτώσεις όπου οι αρμοδιότητες ανήκουν σε διάφορες επιτροπές και στο άρθρο 50. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το άρθρο 50 ακριβώς προβλέπει, όπως ήδη σας ανέφερα, τις δύο υποθέσεις μιας μια έκθεση που εξ ολοκλήρου εμπίπτει σε αρμοδιότητε περισσότερων επιτροπών ή που εν μέρη εμπίπτει σε αρμοδιότητε μια ή δυο ή περισσότερων επιτροπών. Όταν λοιπόν ε, πληρούνται οι όροι που εκτίθενται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 και στο άρθρο 50, η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, εφόσον διαπιστώνει ότι το ζήτημα έχει μείζωνα σημασία, να αποφασίσει ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία με κοινέ συνεδριάσει επιτροπών και μια κοινή ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχοι εισηγητέ συντάσσουν ένα ενιαίο σχέδιο έκθεση, το οποίο θα εξεταστεί και θα ψηφιστεί από τι ενεχόμενε επιτροπέ σε κοινέ συνεδριάσει υπό την κοινή προεδρία των ενδιαφερομένων Προέδρων Επιτροπή οι εμπλεκόμενε επιτροπέ δίνονται να συγκροτήσουν μεικτέ ομάδε εργασία για να προετοιμάσουν τι κοινέ συνεδριάσει και ψηφοφορίε. Άρα, στην ουσία, όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 50, και άρα υπάρχει αίτημα ότι ε, μάλλον διαπιστώνεται ότι το ζήτημα έχει μείζωνα σημασία από τη διάσκεψη των Προέδρων. Στην ουσία, δύο ή περισσότερες επιτροπές, κανονικά συνήθως δύο, ενώνονται σαν να ήταν μία και φτιάχνουν μια έκθεση, έχουν μια διπλή προεδρία, εναλλασσόμενη. Εμεί ήδη το είχαμε αυτό σε εμπειρία με το σχέδιο της Στοκχόλμης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια νέα έκθεση και τις ε, τροπολογίες τις επεξεργαζόμαστε από κοινού. Ποια είναι τώρα τα αιτήματα που μας υποβλήθηκαν. από την διάσκεψη των Πρόεδρων. Τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, η διαδικασία του άρθρου 51 εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας ή μόνο σε πρώτη ανάγνωση. Δεύτερη ερώτηση τα δικαιώματα που συνδέονται με το καθεστώς της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, όπως το δικαίωμα υποβολής τροπολογιών ή πρότασης απορρίψεως στην Ολομέλεια. Μπορούν να ασκούνται μόνο από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές που ενεργούν από κοινού. Τρίτον, σε περίπτωση που πρόκειται για σχέδια κατεξιοδότηση πράξεων εκτελεστικά μέτρα ή που βασίζονται σε νομοθετική ή που έχουν νομοθετικό χαρακτήρα ή προβλέπονται για απονομοθεσία που ήδη έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται παρέμβαση της αρμόδιας επιτροπής. Ισχύει και για αυτή την εκτελεστική λοιπόν φάση η συνεργασία. Αυτά είναι τα τρία ερωτήματα. Μία θέση, μάλλον τρέχω, τρέχω. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Εμείς πρέπει και να αποφασίσουμε αν η απάντηση που πρέπει να δώσουμε θα είναι μόνο μια ερμηνευτική επιστολή ε, με τον κανονισμό κατά αυτόν τον τρόπο, τελεία και παύλα, ή σημαίνει ότι θεωρούμε μάλλον πως είναι σκόπιμο προς χάρη ή για πρακτικούς λόγους να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Να κάνουμε δηλαδή και πρόταση τροποποίηση του κανονισμού. Ο Λένε προτείνει και ένα είδος ε, προσαρτημένου πρωτοκόλου, αλλά στην ουσία πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού. Η διαδικασία προτεινει και ενα ειδος προσαρτημενου πρωτοκολλου αλλα στην λοιπόν, ουσια προκειται για τροποποιηση του κανονισμου η διαδικασια λοιπον του 51 ισχύει μόνο για, το, για την πρώτη ανάγνωση και τα επιχειρήματα υπέρ αυτή τη θέση είναι τρία και τα έχει προτείνει ο συνάδελφος Λένε. Πρώτο επιχείρημα. Μόνο στο άρθρο 51 γίνεται λόγο για μεικτέ επιτροπέ. Γιατί σε πολλά άλλα άρθρα του κανονισμού γίνεται πάντα διάκριση η αρμόδια επί τη ουσία επιτροπή και η αρμόδια για τη γνωμοδότηση επιτροπή. Και εδώ αναφέρονται διάφορα άρθρα, παραθέτονται, όπου, μεταξύ των οποίων το πιο σημαντικό είναι το 108. Αλλά ε, αναφέρεται επίση το άρθρο 66, το 120 κτλ η κοινή θέση του Συμβουλίου πρέπει να ανακοινωθεί στην αρμόδια επιτροπή. Λέει επιτροπή και όχι επιτροπές. Εγώ σας λέω ποια είναι η αποψή μου για να καταλάβετε ποια θα είναι και η τελική μου γνωμοδότηση. Βέβαια εξαρτάται και από τη δική σας άποψη. Κατά την άποψή μου αυτό το επιχείρημα είναι αδύναμο, γιατί το 51 είναι ένα εξαιρετικό άρθρο, ένα έκτακτο άρθρο που λέει ότι αν ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 51, οι δύο επιτροπές λειτουργούν στην ουσία ως μία επιτροπή. Αν αυτό ισχύει λοιπόν σε μία φάση της διαδικασίας, γιατί να μην ισχύει μέχρι τέλους. Και το 108 που μιλάει για ανάθεση στην αρμόδια από ουσίας επιτροπή, στην ουσία αναφέρεται στις ε, αρμόδιες επιτροπές που ορίζει το άρθρο 51 σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω πως αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα άλλο επιχείρημα προτείνει ο ο συνάδελφος λένε είναι πως αυτή η διαδικασία του 51 είναι εξαιρετική, έκτακτη και άρα δεν πρέπει να δοθεί μια εκτεταμένη ερμηνεία αλλά πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο περιορισμένη. Είναι αλήθεια πως πρόκειται για εξαιρετικό κανόνα αλλά αυτοί οι κανόνες ερμηνεύονται στην ουσία με το κυριολεκτικό τους περιεχόμενο και το, το λογικό τους περιεχόμενο. Αν τώρα εμείς λέμε πως δύο επιτροπές να σα δώσω ένα κοινό παράδειγμα. Αν δύο επιχειρήσεις αποφασίσουν από κοινό να χτίσουν ένα κτίριο, φτιάχνουν ε, λοιπόν ένα, μια σύμβαση και λένε ότι η εταιρεία Α θα φτιάξει ε, τι, το μέχρι τον όροφο 20 μαζί με την ε, επιχείρηση Β και μετά τα υπόλοιπα θα τα κάνει μόνη της, είναι δύσκολο μετά να χωριστεί το πράγμα. Όντως είναι έκτακτο και εξαιρετική αυτή η περίπτωση. Όμως είναι εξαιρετική γιατί στην ουσία ε, ορίζει την κοινή εργασία δύο επιτροπών και ε, άλλο επιχείρημα είναι αυτό των ερμηνευτικών δυσκολιών. Το γεγονό ότι γίνεται συνεργασία μεταξύ δύο επιτροπών λέει περιπλέκει ε, το έργο την εργασία του, ιδιαίτερα στην επόμενη φάση, μετά την πρώτη ανάγνωση, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, όταν πρέπει να γίνουν σεβαστές κάποιες προθεσμίες, γίνεται πιο δύσκολο ε, και περίπλοκο. Αυτό το επιχείρημα μάλλον αληθεύει, γιατί δεν έχουμε σχετική εμπειρία, γιατί μέχρι στιγμής οι περιπτώσεις συνεργασίας με βάση το άρθρο 51 ε, ολοκληρώθηκαν στην πρώτη ανάγνωση, άρα δεν χρειάστηκε να περάσουμε σε δεύτερη ανάγνωση. Νομίζω πως μεταξύ της Επιτροπής Γυναικών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών υπάρχουν, υπάρχει μια τέτοια κοινή εργασία, αλλά δεν υπάρχει εμπειρία μέχρι στιγμής για το τι συμβαίνει μετά την πρώτη ανάγνωση. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν ισχύει αυτό το επιχείρημα, ότι είναι αλήθεια δηλαδή ε, δύσκολο να συνεργαστούν δύο επιτροπέ μετά από την πρώτη ανάγνωση, αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε υπάρχει θέμα τροποποίηση του κανονισμού και όχι ερμηνεία, κατά την άποψή μου, γιατί θεωρώ ότι από την άποψη την ερμηνευτική της κατάστασης η απάντηση είναι ότι το άρθρο 51 ισχύει για ολόκληρη τη διαδικασία. Εγώ έτσι το βλέπω. Και βέβαια θα περιμένω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αν υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά την επόμενη φάση, τότε το θέμα είναι η τροποποίηση του κανονισμού. Κατά τη γνώμη μου, το έχω σκεφτεί πολύ. Το έχω σκεφτεί πολύ αυτό το θέμα. διασκέδασα αναλύοντα και ξανααναλύοντας το θέμα. Έχω την εντύπωση λοιπόν πω διαβάζοντας τα άρθρα 49, 50 και 51 από πλευρά του Κοινοβουλίου υπήρξε μια παράληψη. Το άρθρο 51 έχει προετοιμαστεί από μια ομάδα, μια ομάδα, μια ομάδα μάλλον μελέτης που οργανώθηκε από την ε, Προεδρία της Διάσκεψης των Προέδρων και μπορεί κανεί να δει τι εργασίε. Ε, και να τις διαβάσει. Προβλέπετε λοιπόν ότι στην ε, περίπτωση όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο επιτροπών, γίνεται, υπάρχει δυνατότητα να ενοποιηθούν οι εργασίες των δύο επιτροπών. Αυτό είπε εκείνη η ομάδα εργασίας. Όταν στη συνέχεια το Κοινοβούλιο αποφάσισε, ξέχασε αυτό το αίτημα. Μίλησε μόνο για θέματα μεγάλης σημασίας. Εάν πληρούνται, λέει, οι όροι που εκτίθενται στο άρθρο 49 και 50 και πρόκειται για ζητήματα μείζωνος σημασίας, η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αναθέσει κοινή ε, ε, αρμοδιότητα σε δύο επιτροπές. Ωστόσο, το 50 προβλέπει δύο δυνατότητες. Πρώτο, Ένα τμήμα του νομοθετικού κειμένου αφορά αρμοδιότητα μιας επιτροπής, ενώ ένα άλλο τμήμα αφορά αρμοδιότητα άλλης επιτροπής. Και έπειτα απελευρέπει και τη δεύτερη υπόθεση, όπου δεν είναι δυνατή η διάκριση των αρμοδιοτήτων για ολόκληρο το κείμενο. Άρα λοιπόν η ομάδα εργασίας της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών είχε υπογραμμίσει ως προϋπόθεση για την τροποποίηση του κανονισμού είχε υπογραμμίσει την αδυναμία διάκρισης αρμοδιοτήτων για ολόκληρο το κείμενο. Άρα έλεγε λοιπόν ότι και όταν το ζήτημα αυτό έχει μείζωνα σημασία, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με το άρθρο 51. Αυτό λοιπόν εδώ δεν το θυμίζει το 51. Ε, λέει όμως ότι αν πληρούνται οι όροι που εκτίθεται στο άρθρο 50, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να δουλέψουμε από κοινού. Αλλά είναι διαφορετικό το θέμα, γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλουμε να περιορίσουμε στο μέγιστο βαθμό την εφαρμογή του άρθρου 51, σύμφωνα με τη λογική του, δεδομένου ότι μερικώς ε, επικαλύπτει, τις, ε, επικαλύπτονται οι αρμοδιότητες γιατί γίνονται οι γνωμοδοτήσεις των διαφόρων επιτροπών τους ή Θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην περίπτωση όπου δεν γίνεται να υπάρξει διάκριση των αρμοδιοτήτων. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που θέλουμε να τροποποιήσουμε το 51, θα πρέπει να εισάγουμε αυτήν την προπόθεση. Όχι μόνο δηλαδή το ζήτημα να έχει μείζωνα σημασία, αλλά και όταν δεν είναι δυνατή η διάκριση διαφόρων τμήματων αρμοδιότητα στι διάφορε επιτροπέ. Έτσι λοιπόν θα περιοριζόταν και η εφαρμογή του 51. Πιθανότατα, κατά την άποψή μου, δεδομένου ότι αναφέρεται το ζήτημα μείζωνος σημασίας. Και τι σημαίνει τώρα αυτό μεγάλη σημασία. Εύκολα ορίζεται. αν αναφερθεί κανείς στην ε, ρυθμιστική διαδικασία. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να διακριθεί όταν πρόκειται για την εφαρμοστική διαδικασία. Δηλαδή σε εκείνη τη φάση της επιτροπολογίας, όπως την λέγαμε παλιότερα, Ίσως να μην είναι απαραίτητο να ανατρέξει κανείς το άρθρο 51. Όμως πρέπει να το πούμε αυτό ρητά. Αν θέλουμε ωστόσο να βάλουμε μια τροποποίηση, ποιο λέμε τώρα το, σύμφωνα με το 190, 290, δεν θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να επιλέξει μία μόνο επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας όσον αφορά την εποπτεία της εκτέλεσης, της εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Μπορεί να σας φαίνεται ότι έχουμε πολύ μαλλί για ξάσιμο, όπως λέμε και στα Ιταλικά. Ε, πάντως εγώ θα λάβω υπόψη της σα σας για τη σύνταξη ενός τελικού κειμένου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε θερμά για τις εξηγήσεις που μας δώσατε ως προς το πρόβλημα του άρθρου και τις προτάσεις σας για διέξοδο. Εγώ θα πρότεινα να διαγράψουμε τελείως το άρθρο 51. Να παραμερίσουμε τελείως αυτόν το κανόνα. Γιατί η απόφαση για μικτές επιτροπές έγινε από μια θέση αδυναμίας. Και στην πράξη η εμπειρία μας μέχρι τώρα από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ήταν πολύ αρνητική. Είναι πολύ δύσκολο για ένα κοινοβούλιο να δράσει με συνεπή και συνεκτικό τρόπο με τη μέθοδο αυτή. Πάντως αν ξεκολουθήσει να ισχύει το άρθρο 51, συμφωνώ ότι θα πρέπει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Και αν δεσμευτούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις, τις αρμοδιότητες για τις μικτές επιτροπές, θα πρέπει αυτό να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας και να δεσμευόμαστε από την συμφωνία αυτή μεταξύ των Επιτροπών για κοινέ εργασίε. Επίσης, οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατίθενται από κοινού και οποιαδήποτε Επιτροπή αποπειραθεί να αποκλίνει από την κοινή συμφωνία θα πρέπει να στερηθεί αυτή η δυνατότητα, να αναχαιτιστεί αυτή η προσπάθεια. Θα πρέπει να προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να εμένουμε στις ε, αποφάσεις μιας τέτοιας μικτής επιτροπής. και όταν συμπληρώνουμε την απόφαση για την ε, εφαρμογή του 51 θα πρέπει αυτή η διακριτική ευχαίρεια να πορεύει από τη συνδιάσκεψη των Προέδρων. Νομίζω ότι ακριβώ την κατάλληλη στιγμή ήρθε στην ε, συνεδρίαση και ο πρόεδρος της πολιτικής μου ομάδας. Δεν θέλουμε να εμπλέκεται η συνδιάσκεψη των Προέδρων σε ακόμη περισσότερες ε, συγκρούσει αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών. Ιδιαίτερα μετά την έναρξη μιας νομοθετικής διαδικασίας. Ja, im Interesse. Ich möchte mich erstmal zu der Frage äußern, in welcher Form. Ähm, hier Κοιτάξτε, το τι πρέπει να τροποποιήσουμε και πώς είναι το θέμα. Αν θα τροποποιηθεί ο κανονισμός δηλαδή και δεν περιοριστούμε απλώς σε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές που να κάνουν παραπομπή σε κάποιο άρθρο του. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε στη διά, να το αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Μάλλον πρέπει να τροποποιήσουμε τον κανονισμό, έτσι θα είναι τα πράγματα σαφέστερα. Δεύτερον, αν η τροποποίηση θα αφορά ολόκληρη τη διαδικασία ή μόνο την πρώτη ανάγνωση, συμφωνώ με τη νομική σας γνωμοδότηση. Στο σύνολο της, το σύνολο της διαδικασίας να αφορά η αλλαγή. Τα επιχειρήματά σας ήταν πολύ πιστικά και οποιαδήποτε άλλη απόφαση δεν θα είχε νόημα, διότι μια νομοθετική διαδικα... η νομοθετική διαδικασία έχει διάφορες φάσεις και όχι μόνο την πρώτη ανάγνωση δεν θα είχε νόημα λοιπόν να τροποποιήσουμε τον κανονισμό για μία από τις φάσεις αυτές. Όσο για τα υπόλοιπα ερωτήματα, το δεύτερο και το τρίτο ιδιαίτερα, εκεί δεν θα απαντήσω γιατί δεν είμαι αρκετά, δεν με ενδιαφέρουν αρκετά. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Αν τροποποιηθεί ο κανονισμός για αποσαφήνιση δηλαδή, τότε επειδή είμαι καινούργια στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να πω ότι η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών επίσης επηρεάζεται από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες και οι βουλευτές που δεν παρίστανται εκεί δεν μπορούν εύκολα να καταλάβουν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Ο Γουίδων Παρακολουθήσαμε μια πραγματικά καταπληκτική διάλεξη για το Ιταλικό Δημόσιο Δίκαιο και ήταν τόσο καταπληκτική αυτή η διάλεξη που μας κάνατε κύριε Πρόεδρε που κάπως ε, μπερδευτήκαμε στη συζήτηση. Υπάρχει ένα θεμελιώδη ζήτημα εδώ που καλούμαστε να επιλύσουμε δεν έχουμε πρόβλημα στην πρώτη ανάγνωση μιας νομοθετικής διαδικασίας. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση ισχύουν και λειτουργούν και οι δύο εμπλεκόμενες επιτροπές. Το πρόβλημα ανακύπτει στη δεύτερη ανάγνωση, σε περίπτωση που θα φτάσουμε σε φάση δεύτερης ανάγνωσης. Γιατί, όπως είπε και ο Πρόεδρος, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει δείξει ότι τα πράγματα διαθετούνται ήδη στην πρώτη ανάγνωση. Σε περίπτωση όμως που φτάσουμε και σε στάδιο δεύτερης ανάγνωσης, το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι διαδικαστικό. Τα προβλήματά μας είναι διαδικαστικά, θα είναι θέματα προθεσμιών, η πίεση χρόνου για να διαμορφώσουμε κάποιες συμφωνίες. Δεν αμφισβητείται εδώ αν και οι δύο επιτροπές θα πρέπει να συμμετέχουν στην τελική απόφαση μιας νομοθετικής διαδικασίας. Γιατί όλοι ως προς αυτό συμφωνούμε ότι η νομοθετική διαδικασία είναι ενιαία Οπότε τη στιγμή που λαμβάνεται η τελική απόφαση, η οριστική απόφαση, εμπλέκονται και οι δύο επιτροπέ. Δεν είναι στη στιγμή τη τελική απόφαση που θα καταργηθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Ω προ την ουσία, συμφωνούμε ότι εμπλέκονται μέχρι τέλου οι επιτροπέ. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε ίσω μία νομοθετική διάταξη, ένα άρθρο που θα διέπει τα διαδικαστικά προβλήματα της δεύτερης ανάγνωσης για τις ε, νομοθετικές διαδικασίες. Ώστε να αποφύγουμε να λαμβάνει συνεχώς ε, αποφάσεις στη συνδιάσκεψη των Προέδρων. Επειδή υπάρχει μια διαδικασία που περικόπτει τις προθεσμίες ή υποχρεώνει τις Επιτροπές να συνεργαστούν με διαφορετική μεθοδολογία από τη συνηθισμένη που είναι, είναι αυτή που ισχύει όταν έχουμε μόνο μία επιτροπή. Θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοια συνεχή εμπλοκή της συνδιάσκεψης των Προέδρων. Δεν βλέπω άλλο να έχεις δει το, το, λόγο. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να προχωρήσω και να συντάξω μια έκθεση αυτή καθ' αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα τους δικούς σας που για την ώρα α, θεωρώ ότι είναι η εξή. Προσανατολιζόμαστε προ τροποποίηση του κανονισμού και όχι προ ερμηνευτική επιστολή. Νομίζω πω αυτό είναι η άποψη όλων. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή η διαδικασία να ισχύει σε ολόκληρη την νομοθετική διαδικασία και όχι μόνο σε μία φάση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της δεύτερης φάσης και της τρίτης ώστε να επαληθεύσουμε όλες τις προθεσμίες και τα λοιπά, θα το κάνουμε. Τώρα, δεν βρήκα καμιά αντίρρηση όσον αφορά αυτή την πρόταση που νομίζω ότι είναι σημαντική επίσης, δηλαδή να εισαχθεί στο άρθρο 51 πέρα από την προϋπόθεση της σημασίας του ζητήματος και η προϋπόθεση της μη διακριτής αρμοδιότητας δηλαδή για ολόκληρη την έκθεση. Αυτή είναι η δυσκολία που οδηγεί στο να ανατεθεί σε δύο επιτροπές μια έκθεση και όχι σε ορμονομία. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα διάκριση των αρμοδιοτήτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτή να είναι μια ελάχιστη προπόθεση για την εφαρμογή του 51. Θα προετοιμάσω λοιπόν την έκθεση. Ε, τώρα θα πάμε έτσι και αλλιώς για Γενάρη. Θα κάνετε εσεί τι παρατηρήσει σα, τι τροπολογίε σα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο προσανατολισμό είναι αυτό. Δηλαδή μια μικρή τροποποίηση του κανονισμού. Σα ευχαριστώ. Και τώρα Περνάμε στο τελευταίο σημείο που προβλέπεται για σήμερα και είναι μια συζήτηση για τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου. Στην πράξη δεν πρόκειται για όλα τα πορίσματα, όλα τα συμπεράσματα, αλλά για εκείνο το κομμάτι των συμπερασμάτων που αφορούν την συνταγματική διάσταση, δηλαδή το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και της σχετικής task force. Τώρα, δεν ξέρω πώ να παρουσιάσω τώρα αυτή τη συζήτηση. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό θέμα θα ήταν να Το πιο σοβαρό θα ήταν να το διαβάσετε το συμπέρασμα. Τα έχετε δει, το έχετε δει το επίσημο κείμενο. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το συμπέρασμα που ήδη γνωρίζετε. Ίσως ο συνάδελφος Νταβ που ζήτησε κιόλα να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη αυτό εδώ το θέμα να ήθελε να μας προ... ξεκινήσει τη συζήτηση. Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνείτε να γίνει μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων καταρχήν γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Επιτροπή μας αλλά και για το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Οι αλλαγές της συνθήκης θα μπορούσαν, για μένα τουλάχιστον, να αποτύχουν και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τι θα πούμε, πώς θα απαντήσουμε στα συμπεράσματα αυτά του Συμβουλίου. Φαίνεται ότι προτείνουν αλλαγή του άρθρου 122, εδάφιο 2 ώστε ώστε να αλλάξει το νόημά του και να επιτρέπεται η εφαρμογή ενός προσωρινού μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων σε μόνιμο Υπάρχουν βέβαια μεγάλες δομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και αυτό θα μπορούσε και θα μπορούσε κανείς να πει ότι σε όλες εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν μπορούν να ελεγχθούν από μεμονωμένα κράτη-μέλη μπορεί να δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Ότι η κατάσταση έχει καταναντήσει χρόνια δηλαδή και όχι εξαιρετική. Πρόκειται βέβαια για σημαντική αλλαγή στην, ε, στο νόημα, στην ερμηνεία του άρθρου και δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να συνδυαστεί με το 125 όπου ρητά υπάρχει απαγόρευση της ρήτρα των προσωρινών εξαιρέσεων bailout. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε αν το αίτημα αυτό για μία αλλαγή της συνθήκης είναι αποδεκτό από εμά ή όχι. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων γίνεται για να αντιμετωπιστεί κάποιο έλλειμμα, κάποια έλλειψη κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κράτος μέλος ιδίως όσον αφορά το χρέος του, τότε η αλλαγή αυτή θα ήταν τόσο σημαντική ώστε θα σήμαινε υποχρεωτικά και μεταφορά αρμοδιοτήτων. Αν όντως έτσι συμβαίνει τότε το 48.6 που προβλέπει την απλοποιημένη διαδικασία αλλαγής της συνθήκης δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πρέπει σε αυτή την περίπτωση να περιμένουμε για να δούμε τι ακριβώς προτείνουν πριν γνωμοδοτήσουμε. Επίσης όμως μου φαίνεται ότι αν γίνει αυτή η αλλαγή τότε η αλλαγή δεν είναι επαρκής απάντηση στο πρόβλημα της κατάργησης των ρυθμίσεων του Μάστριχτ για τη ρύθμιση των προβλημάτων που δημιούργησε η Νομισματική Ένωση και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ή οι πολίτες δεν πρόκειται να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους. εκτός εάν υπάρξει μια πραγματική κοινή ομοσπονδιακή διακυβέρνηση. Προφανώς δεν πρόκειται να εγκριθεί κάτι τέτοιο τώρα, αλλά λογικό θα ήταν νομίζω εμείς ως Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία ως προς την ε, απλοποιημένη και φαινομενικά ε, απλή αυτή η αλλαγή μεταρρύθμιση της συνθήκης ώστε οι περαιτέρω ποιοτικέ αλλαγές που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση της κρίσης να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Εάν το Συμβούλιο θέλει απλώς να συγκεντρώσει, να κάνει ένα συντονισμό των ε, εθνικών οικονομικών προγραμμάτων αλλά δεν εφαρμόσει μια κοινή ομοσπονδιακή πολιτική τότε νομίζω ότι απράττει τεράστιο λάθος. Εν μέρη διότι ενισχυμένος συντονισμός ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να λειτουργήσει στο μέλλον όπως δεν λειτουργήσε ούτε στο παρελθόν. Αλλά επίσης και διότι θα θεωρηθεί ως δημοκρατικός απαράδεκτο βήμα. Τέλος, αν θέλουμε, και συμφωνούμε νομίζω από αυτό ότι θέλουμε, να ενδυναμώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, διαχείριση, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι και για να βελτιωθεί η δημοκρατική νομιμότητα των θεσμών της Ένωσης, των θεσμικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και το Κοινοβούλιο. Γνωρίζετε ότι οι προτάσεις μου για την εκλογική μεταρρύθμιση των ευρωεκλογών προβλέπουν και αυτές αλλαγή στη συνθήκη. Και η απάντηση που θα δώσουμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια αναφορά, μια παραπομπή και στο θέμα αυτό του κατά πόσον θα έπρεπε να βελτιωθεί η δημοκρατική νομιμότητα του Κοινοβουλίου εφόσον επαναλαμβάνω θέλουμε να επιβάλλουμε στον φορολογούμενο και τη φορολογούμενη μια ενισχυμένη μορφή οικονομικής διακυβέρνησης που να συμπεριλαμβάνει και ένα μόνιμο μέσο μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Νομίζω αυτά είναι τα σοβαρά ερωτήματα που ως Επιτροπή πρέπει να συζητήσουμε και μάλιστα διεξοδικά και πρέπει να μας πληροφορήσει και η Κομισιόν και ο πρόεδρος Βαν Ρόμπουι. Να μας πούν δηλαδή τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν πριν μπορέσουμε να αποφασίσουμε την γνωμοδότηση που θα δώσουμε στο Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια δηλαδή. Ευχαριστούμε. κύριε Τάφ. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Μένες Δεβίγκο. Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν γύρω από την συνταγματική συνθήκη είχε συγκροτηθεί και μία ομάδα εργασίας για την εξέταση και την ανάλυση των αλλαγών που θα μπορούσαμε να επιφέρουμε στη συνθήκη από οικονομική άποψη. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν και πολύ ε, λαμπρό, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία. Και η μοναδική μεταρρύθμιση που εγκρίναμε τότε ήταν να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. Κατόπιν έλαβε χώρα η διακυβερνητική συνδιάσκεψη, ήρθαν οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και είπαν οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις συντονίζουν μεταξύ τους τις οικονομικές πολιτικές στο πλαίσιο της Ένωσης. Είναι σημαντική αυτή η διαφορά στη διατύπωση. Στην εισαγωγή που μας έκανε ο κύριος Ντάφα, δεν ανέφερε την έλλειψη, την πεντελή έλλειψη πολιτικής βούλησης για οποιαδήποτε αλλαγή. Στο μεταξύ ενέσκυψε η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση και φυσικά τα πράγματα επιταχύνθηκαν ραγδαία τον τελευταίο καιρό. Αρκεί να ρίξει κανεί μια ματιά στις οδηγίες και τους κανονισμούς σε ό,τι αφορά τις Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας σε τραπεζικά θέματα ασφαλίσεων, την Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου έγιναν πολύ εντυπωσιακές αλλαγές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης ε, που διαπιστώσαμε τότε στη συνθήκη έδωσε τη θέση της σε μια κατάσταση ανάγκης που επιτάχυνε τα πράγματα και που Μα οδήγησε στην πέρασμα ότι η προηγούμενη κατάσταση δεν παρκούσε για να αντιμετωπιστούν τα πρόσφατα προβλήματα. Η κατάσταση άλλαξε πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Βλέπουμε τις αναδυόμενες οικονομίες, δεν ξέρω αν επέδρασε και αυτές. Πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε η Κίνα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Οπότε, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αλλαγής και στο νομοθετικό ζήτημα και στην τροποποίηση, την αλλαγή των συνθηκών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι και πολύ σαφή τα πράγματα. Ε, η δική μου πολιτική ερμηνεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Κορυφής είναι ότι ανατέθηκε στον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Βαν Ρομπαϊ, η εντολή να εξετάσει τι θα μπορούσε να προτείνει και μόνο ένα συγκεκριμένο πράγμα υπάρχει στα συμπεράσματα. Η βούληση, η δεδηλωμένη βούληση να δοθεί μια νομική βάση και να κλειδωθεί νομικά αυτός ο μηχανισμός διάσωσης. Δεν έχω καμία αμφιβολία για τους λόγους που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Και ένα σχολαστικό στεγματικό δικαστήριο ίσως κρίνει ότι δεν υπάρχει επαρκή νομική βάση στο άρθρο 122 για την σύσταση ε, του μηχανισμού αυτοδιάσωσης με μόνιμο χαρακτήρα. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε τα πιθανά προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι δεν επιλύεται έτσι η κατάσταση. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο τμήμα, ένα μεμονωμένο τμήμα της κατάστασης. Και ο κύριος το είπε πολύ γλαφυρά είπε ότι ενώ είμαστε στη θάλασσα τότε προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις ε, σωσίβιες λέμβους για να γλιτώσουμε. Αλλά οι σωσίβιες λέμβοι δεν είναι ολόκληρο το πλοίο, είναι ένα μικρό τμήμα του μεγάλου σκάφους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το πώς θα εφαρμοστούν οι προτάσεις Βανερόμπο για άλλα θέματα και αν θα γενικευτούν. Δεν ξέρω τι θα γινόταν με μια πιο φιλόδοξη συζητήσιμη πρόταση που θα πρόβλεπε την αυτόματη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για το έλλειμμα εκ μέρους ενός κράτους ή της πρότασης υποβολής των κρατικών προϋπολογισμών πριν τη συζήτησή τους στα Εθνικά Κοινοβούλια για να και να κρίνουν οι ευρωπαϊκές αρχές κατά πόσο αυτοί οι κρατικοί προϋπολογισμοί συμφωνούσαν και ευθυγραμμίζονταν με τους σκοπούς της ε, συνθήκης ή της διατάξης της συνθήκης. Πάντως έχω την αίσθηση ότι με της συνθήκης είναι αυτό το συγκεκριμένο μεμονωμένο τμήμα ή τίποτα. Αν όμως ισχύει κάτι τέτοιο, εγώ πραγματικά θα προβληματιζόμουν πολύ σοβαρά, γιατί πιστεύω ότι το να δώσουμε μια μόνιμη νομική βάση και μόνιμο χαρακτήρα στο μηχανισμό διάσωσης μπορεί να επιλύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά δεν αγγίζει καθόλου κάτι που πραγματικά ε, υποχρεώνει σε αλλαγή μετά την φυσική φθορά της συνθήκης του Μάστριχ μετά από μία εικοσαετία εφαρμογή. Γιατί σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πια θέλει διεκδικεί μεγαλύτερη ισχύ στα οικονομικά θέματα. Εμένα δεν με προβληματίζουν οι όροι οικονομική διαχείριση, οικονομική διακυβέρνηση. Νομίζω θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι ε, εμπλεκόμαστε τώρα στη συζήτηση ενός πολύ αποσπασματικού κανόνα με μια πολύ περιορισμένη μεταρρυθμίση που δεν θα περνάει από μια νέα ε, συνέλευση συντακτική. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, λένε ότι αυτό θα γίνει για να ενταχθεί σε ένα πακέτο, ίσως στα πλαίσια της επόμενης διεύρυνσης με την ένταξη της Κροατίας. Και όταν μιλούμε για την επικύρωση του 2013, μέχρι το 2013 όμως, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει στον πολιτικό ρόλο του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πιστεύω ότι αυτή η πρόταση που μπορεί να είναι απαραίτητη από νομική άποψη και αντιλαμβάνουμε τις δυσκολίες που μπορεί να έχει συγκεκριμένο κράτο μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι επαρκή αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί είναι πολύ βραχία, πολύ περιορισμένη. Και θα ήταν σκόπιμο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η ομάδα του Βαν να εμβαθύνει στο θέμα αυτό και να υποβάλει πιο μεγαλεπίβολε προτάσει, πιο φιλόδοξε και ευρύτερε. Εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε φυσικά πρόθυμοι να συνεργαστούμε ήδη από τώρα, ήδη από αυτή τη φάση και πιστεύω ότι αν εγκριθούν πραγματικά μεγάλε επίβολε μεταρρυθμίσει, μεγάλε ευέλειε, ίσω το σκόπιμο να γίνει αυτό στο πλαίσιο μια νέα συντακτική συνέλευση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αναλύουμε και να επιλύουμε όλα αυτά τα θέματα τα σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης ερήμην μίας, ε, στο περιθώριο μιας ε, συνέλευσης, χωρίς μια τέτοια συνταγματική συνέλευση γιατί μιλούμε για νομιμοποίηση. Εγώ ήμουν κατά τη μεθόδου τη συνταγματική συνέλευση για συγκεκριμένε, περιορισμένε και μεμονωμένες μεταρρυθμίσει. Αλλά αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη, κατά πάσα πιθανότητα και απορρέει και από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, είναι μια πιο ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση. Οπότε το μήνυμα προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ήταν σκεφτείτε και αναλύσετε μήπω αυτό το περιορισμένο ε, μεμονωμένο τμήμα νομικό θέμα της νομικής βάσης για το άρθρο 122 μήπως χρήζει πιο ευρυθούς και εις βάθος συζήτησης για την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Και από την άποψη αυτή κύριε Πρόεδρε πιστεύω ότι ο ρόλος μας θα ήταν και πάλι να γίνουμε κινητήριο κινητήριος μοχλός και να προωθήσουμε πιο βαθίε μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το μήνυμά μας και αυτή είναι η αποστολή μας, να στείλουμε αυτό το μήνυμα και φυσικά να δούμε πώς θα δρομολογηθεί στου επόμενου μήνε αυτό το θέμα. Ο στήμα τη εντολή που έχει ο πρόεδρο Βαν Ρόμπαϊ είναι να συζητήσει με τα κράτη-μέλη, αλλά φαντάζομαι και με τα υπόλοιπα κοινοτικά θεσμικά όργανα, για να δούμε ποια είναι κατά τη γνώμη μα το σωστό περιεχόμενο αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και με βάση όσα λέμε εδώ, καλό θα ήταν να συζητήσουμε το θέμα και με τον πρόεδρο μας, τον κύριο Μπούζεκ, προκειμένου να διαβάσουμε μέσω εκείνου τους στόχους μας και τις παρατηρήσεις μας για τις ανάγκες της Ένωσης. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια που είχατε την ε, ιδέα να συγκαλέσετε αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Ε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σα. Ο κύριος Φερχόφστατ ζήτησε να μιλήσει. Έχετε το λόγο. Χωρί μικρόφωνο μιλητής. Ε, Κοιτάξτε, κανονικά τα θέματα αυτά συζητούνται στην Οικονομική Επιτροπή όπου προβλέπονται όχι λιγότεροι από έξι εισηγητέ για την ουσία του θέματος. Και πρέπει καταρχάς να πούμε και να διαπιστώσουμε ότι οι αντιδράσεις για όλη τη δέσμη και των συμπερασμάτων υπήρξαν ε, όχι και πολύ ομόφωνες. Εγώ Άκουσα τι είπε ο κύριος Τρισέ, ο οποίος όπως ξέρετε είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο οποίος την Παρασκευή στον τύπο, μία εβδομάδα μετά τη διάσκεψη λοιπόν, επανέλαβε τους φόβους του για την αποφασισμένη δέσμη. Είπε ότι δεν αρκεί όπως έλεγε και ο κύριος Μέντες Δεβίγο. Δεν αρκεί και χρειάζεται κάποιος μηχανισμός ή κάποιοι μηχανισμοί πολύ πιστικότεροι και πρέπει να μπορέσουμε να πάμε πολύ μακρύτερα από αυτά που αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του κυρίου Τρισέ νομίζω εννοούν ότι οι μηχανισμοί που αποφασίζονται και από το διορθωτικό τμήμα και από το αποτρεπτικό τμήμα δεν αλλάζουν το πρόβλημα, δεν λύνουν το πρόβλημα γιατί ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να αρχίσει να τίθεται σε λειτουργία μόνο από το Συμβούλιο στο 121 και 126 της συνθήκης και στις δύο περιπτώσεις 121 για την οικονομική πολιτική και στο 126 για το σύμφωνο σταθερότητας για να μην υπάρχουν υπερβολικά υψηλά ελλείμματα και στις δύο περιπτώσεις το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να αρχίζει να θέτει σε λειτουργία τη διαδικασία ή το μηχανισμό και τα τέλη Σεπτεμβρίου, 29 Σεπτεμβρίου αν δεν με, η Task Force, των οποίων τα συμπεράσματα τα δέχτηκε και το Συμβούλιο, σε αυτά τα δύο άρθρα βασίζονται. Δεν γίνεται αλλιώ αφού η συνθήκη αυτή είναι. Δεν αλλάζουν τα συμπεράσματα ενός Συμβουλίου τη συνθήκη. Βασίζονται λοιπόν σε ένα, μιλάνε για ένα μηχανισμό όπου πρέπει με ενισχυμένη πλειοψηφία να διαπιστωθεί πρώτα ότι υπάρχει πρόβλημα για να μπορέσει να αρχίσει να, εφαρα... να λειτουργεί ο μηχανισμός. Και άρα χρειάζεται καταρχάς μια πολιτική απόφαση με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αν μια χώρα δηλαδή κατορθώσει να δημιουργήσει μειοψηφία που να εμποδίζει να παγώνει τα πράγματα, σταματάνε τα πάντα. Ε, θυμάμαι μια περίπτωση που η Γερμανία δεν ήθελε σε ορισμένε περιπτώσει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το Σύμφωνο Σταθερότητα, δεν εφαρμόστηκαν. Το 5 έγινε αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι οι δέσμοι αυτοί είναι μεν πρόοδος, υπάρχουν σίγουρα βελτιώσεις. Αλλά παραμένει το βασικό πρόβλημα ότι δεν πρόκειται πραγματικά για μηχανισμό ούτε κάνει μη αυτόματο αφού χρειάζεται προποηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου. Και άρα Βέβαια δεν μπορούσε να αποφασιστεί τίποτε διαφορετικό αφού αυτό προβλέπει συνθήκε στο 126 κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, ότι δηλαδή η αλλαγή του 122 θα μπορούσε να δώσει μια πιο σταθερή και μόνιμη βάση σε έναν τέτοιο μηχανισμό παρέμβασης και νομίζω πρόεδρε ότι όλοι βλέπουμε ότι και οι αγορές μπορεί μεν να βελτίωσαν την κατάστασή τους και για την Ελλάδα και για την Πορτογαλία αλλά σήμερα μετά τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ελλάδα ξανά πέσαν οι τιμές, στην Ιρλανδία ξανανέβηκαν, στην Πορτογαλία επίσης, ε, δηλαδή παραμένουν τα πράγματα φλού. Αυτό εννοώ. Όλη αυτή η συζήτηση ενδιαφέρει και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τι πρέπει λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε ως θέση. Κάποτε θα χρειαστεί, δεν ξέρω πότε, το Δεκέμβριο φαντάζομαι ή λίγες εβδομάδες μετά, θα χρειαστεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει το 48-6 Δηλαδή μία απλή αναθεώρηση και όχι μεταρρύθμιση. Τι θα πούμε εμείς όμως. Χωρίς συνεδρίαση και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου δεν υπάρχει αλλαγή της συνθήκης. Και εμείς έχουμε κάποιο ρόλο αλλά δεν είναι ο ίδιος. Για πρώτη φορά θα έχουμε και εμείς ένα ρόλο λοιπόν και πρέπει να γνωρίζουμε από τι εξαρτάται η θέση που θα λάβουμε. Καταρχήν τι είναι αυτή η αλλαγή που προτείνεται. Δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε σήμερα αφού δεν έχουμε το ίδιο το κείμενο για την αλλαγή του 122 για να μπορέσουμε να κρίνουμε τι σημασία έχει η αλλαγή αυτή, αν είναι βαθιά ή όχι. Και δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει επίσης να περιμένουμε τι θα μας πει η Οικονομική Επιτροπή, διότι είναι πιθανό να μας προτείνουν και άλλες αλλαγές της συνθήκης. Ή μίλησα πριν για τον μηχανισμό που προτείνεται τώρα, που τον περιορίζουν τα 122 και 126, αλλά μπορεί να υπάρχουν, να παίζουν εδώ και τα άρθρα που αφορούν την νομισματική πολιτική. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι απαιτείται πολιτική απόφαση του Συμβουλίου ενώ οι αγορές αυτόματα εφαρμόζουν τις αλλαγές. Επομένως, ο στόχος μας πρέπει να είναι η ενωσιοποίηση ή κοινοτικοποίηση του μηχανισμού. Ε, για να υπάρξει αυτό χρειάζεται αλλαγή της συνθήκης, χρειάζεται άλλο άρθρο, καινούριο. Αν θα είναι 121, 126 δεν ξέρω, μπορεί να αφορά μόνο την Ευρωζώνη ή τα νομισματικά. Πρέπει όμως πρώτα να δούμε τι θα πούν οι δήμονές μας στην Επιτροπή Εικόν. Αν συμφωνούν ότι πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω από την πρόταση του Συμβουλίου ή αν μπορούμε να δεχτούμε την πρόταση ως έχει. Τελικά όμως η ουσία είναι ότι πρέπει να περιμένουμε την πρόταση που θα μας κάνει το ίδιο το Συμβούλιο για να δούμε πώς ακριβώς αλλάζει τα πράγματα για το 122. Και καταλήγω κύριε Πρόεδρε, φυσικά είναι προφανές ότι δεν μπορούν να μας πούνε εμάς στο Κοινοβούλιο ότι θα αλλάξουμε ένα μόνο άρθρο στη συνθήκη αλλά απαγορεύεται να αλλαγεί και δεύτερο. Αυτό είναι η τακτική του Συμβουλίου, να αλλάξει ένα άρθρο για να μπορέσει να εφαρμοστεί το σύστημα που προτείνουν, ενώ η Γερμανία επιμένει να περιοριστούμε ακριβώς αυτό, στο 122 μόνο. Εμείς μπορούμε να υποφεληθούμε για να αλλάξουμε και άλλα άρθρα. Να πούμε δηλαδή ότι για να υπάρξει όντως αυτός ο μηχανισμός χρειάζεται αλλαγή και άλλο άρθρο. Το ίδιο το επιχείρημα του Συμβουλίου δηλαδή που χρησιμοποιεί σήμερα το Συμβούλιο για να αλλάξει η συνθήκη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς για να λειτουργήσει καλύτερα ο μηχανισμός. Πρώτα όμως πρέπει να έχουμε το κείμενο της αλλαγής του 122 που προτείνει το Συμβούλιο και μετά να δούμε τι θα πούνε οι δικοί μας στην Επιτροπή Εικόν. Να δούμε αν θεωρούν ότι αρκεί αυτή η πρόταση ή πρέπει να πούμε και τίποτε άλλο. Σα ευχαριστώ. Το λόγο ζήτησε ο κύριο Γουαλτιέρη. Σα ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι διανύουμε μια πολύ κρίσιμη στιγμή όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο, να καθορίσει μια στρατηγική, να προσδιορίσει σαφείς στόχους Προφανώ στη συνέχεια όταν θα υπάρξει πρόταση όπως έλεγε και ο Φερχόφστατ αλλά σίγουρα εμείς ε, θα πρέπει να προετοιμαστούμε γέρο, διότι η φύση της πρότασης αυτής, της τροποποίηση δηλαδή το 122 μπορεί κανεί να την ε, υποψιαστεί. Όπω έλεγε ο Φερχόφστατ, η προεπόπειρα θα είναι να γίνει όσο γίνεται πιο μικρή μεταρρύθμιση που να επιτρέπει την μόνιμη ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού ύφεση ή κρίσης που θα ξεπεράσει έτσι τη μεγάλη θεσμική δημιουργικότητα που θα μπορούσε να επιτρέψει να ξεπεραστεί το 122 δύο τους περασμένους μήνες. Συμφωνώ απόλυτα με την κρίση των υπολείπων συναδέλφων ότι δηλαδή ε, γίνεται πόπειρα να κατευθούμε σε ακατάλληλο πορεία Να δημιουργηθούν δηλαδή μηχανισμοί και δομέ που όλα ένα και περισσότερο θα ξεπερνούν, θα παρακάμπτουν την κοινοτική μέθοδο, διάφορε ε, οργανισμοί, επιοργανισμών κτλ. Πάντω σίγουρα δεν μα πείθει αυτή η γραμμή. Το θέμα είναι ποια είναι η τακτική, ποια είναι η πιο αποτελεσματική η στρατηγική που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε μια κοινή συζήτηση με του συναδέλφου τη Οικονομική Επιτροπή, ΑΦΚΟ, ΕΚΟΝ, για να συζητήσουμε από κοινού συνταγματικά και οικονομικά αυτά τα θέματα του 122, 126, 121 και να αρχίσουμε να εντοπίζουμε αρκε, ακριβώς τι αντισταθμίσματα θα είναι ρεαλιστικά αλλά και ταυτόχρονα φιλόδοξα ώστε το κοινοβούλιο να μην μείνει στην άκρη και να μην παρακαμφθεί με βάση μια τέτοια απλοποιημένη τροποποίηση. Να έχουμε δηλαδή ουσιαστικά αντισταθμίσματα Ρεαλιστικά, ωστόσο. Βεβαίω δεν θα μπορούμε τώρα στην ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει να αρχίσουμε να εντοπίζουμε κάποια στοιχεία. Ήδη αναφέρθηκαν κάποια από αυτά. Εγώ λοιπόν σε σχέση με τα όσα έλεγε ο Άντριου Νταφ καταλαβαίνω την σημασία του θέματος της δημοκρατικής νομιμότητας αλλά ίσως εγώ θα έμενα στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα και για μένα το πιο σημαντικό είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού διαχείρισης της κρίσης. Δηλαδή, ναι, μπορούν να αλλάξουν και άλλα άρθρα, αλλά υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι να αλλάξει το 122. Έπειτα βεβαίως υπάρχουν τα άλλα θέματα τα οποία ε, θα θίξει, ε, μάλλον έθιξε ο Βερχόσταφ και ίσως από αυτά θα ξεκινούσε μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Ίσως ήταν πιο λογική η συνέλευση. Υπάρχουν πάντως και άλλα θέματα τα οποία συζητώνται ταυτόχρονα μέσα στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο, όπου το θέμα είναι ο προπολογισμό τη γραμμή 11 να περιλάβει και κάποια στοιχεία όπω οι ήδη πόροι ε, μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Συζητείται και αυτό. Να συμμετέχει λοιπόν η ΕΚΟΝ, η ΑΦΚΟ, οι πολιτικέ ομάδε, γιατί είναι ένα θέμα εξόχω πολιτικό, πολιτική φύση, και να προετοιμαστούμε για μια διαπραγμάτευση την οποία θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω, έχοντα ήδη στην τσέπη μας κατοχυρωμένα δηλαδή κάποια στοιχεία αντισταθμίσματα που θα θέσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τέιν. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ρεαλιστική η απόφαση του Συμβουλίου. Ίσως θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες λύσεις αλλά για κάτι τέτοιο θα πρέπει να τροποποιήσουμε άρδιν τη συνθήκη. Και άρα θα χρειαστούν δημοψηφίσματα σε πολλέ χώρε. Και είδαμε τι συνέβη με άλλε μεταρρυθμίσει τη συνθήκη και τι έγινε με τα δημοψηφίσματα. Πιστεύω ότι αποκλείεται να έχουμε τέτοιε μεταρρυθμίσει μέχρι το 2013, που είναι και η προθεσμία εκπνοή του σχεδίου διάσωση. Οπότε ανακύπτει το ζήτημα μήπως είναι σκόπιμες πιο περιορισμένες μεταρρυθμίσεις της συνθήκης, γιατί αυτό το σχέδιο διάσωσης ουσιαστικά θεσπίστηκε εις βάρος των ε, Γερμανών φορολογουμένων και έχουν ασκηθεί πολλές προσφυγές στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα δημιουργηθούν προβλήματα με τη λύση αυτή. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο δεν μπορεί να συνεχίσει με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάνει ειδήμων στα συνταγματικά ζητήματα για να δει ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η πορεία μακροπρόθεσμα. Βέβαια, καλλιοπέντε και στο χέρι σκέφτονται πολύ, γι' αυτό ίσω είναι σκόπιμε περιορισμένε μεταρρυθμίσει τώρα από το να περιμένουμε το 2013. Προ το παρόν και μέχρι το 2013, άλλη λύση μεγαλύτερη εμβέλεια δεν είναι εφικτή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για πιο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση. Δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία για τέτοια φιλόδοξη πριν την κρίση και ούτε καν τώρα μεσούσε της κρίσης. Ευχαριστώ κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο κανείς να προετοιμαστεί για μια συζήτηση όταν ε, τροποποιείται τελευταία στιγμή μερίσια διάταξη. Η πρόταση για την αλλαγή του άρθρου 122, το συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής ε, πολιτικής, αφορά μόνο τις χώρες της Ευρωζώνης. Τέτοιου όμως αλλαγές πολύ συχνά ακολουθούν τη δική τους πορεία. Διαρωτώ με αν σκεφτήκαν τα μέλη της Επιτροπής μας ότι αυτό το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης μπορεί να επεκταθεί και σε, ζώνες, σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Γιατί απότερο σκοπό. των, ε, με, με την προπόθεση ότι απότερο σκοπό όλων των χωρών τη Ένωση είναι να γίνουν κάποια στιγμή μέλη τη Ευρωζώνης. Κάτι τέτοιο όμω προϋποθέτει εκχώρηση ε, κυριαρχία σε οικονομικά θέματα που προϋποθέτει διεξαγωγή δημοψηφίσματος στο ε, Ενωμένο Βασίλειο. Βέβαια, αυτό είναι θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου, αν θα κάνει δημοψήφισμα και θα συμφωνήσει με κάτι τέτοιο και όχι της Επιτροπής. Ο κύριος Μορέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο θεμάτων εδώ. Το ένα είναι τι μέτρα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει το πρόβλημα και το έλλειμμα της οικονομικής διακυβέρνησης που αναδείχθηκε από την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Και επίσης να δούμε τι τροποποίησεις ε, είναι απαραίτητες ε, στη συνθήκη για να αρθούν τα εμπόδια σε αυτή την πολιτική μεταρρύθμιση. Κάτι που αφορά τη δική μας Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το ανακοινωθέν του και τα συμπεράσματά του Μιλάει για ανάγκη τροποποίησης μόνο του άρθρου 122 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δοθεί και μια συνταγματική νομική βάση σε έναν μόνιμο μηχανισμό οικονομικής χρηματοπιστωτικής διάσωσης των χωρών. Και αυτό είναι, ήταν μια ανησυχία της Γερμανίας περισσότερο και πρωτοβουλία της Γερμανίας που ε, πηγάζει από το φόβο της Γερμανίας να απορριφθεί από το ε, Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο το, η νομική βάση της, ε, ε, του μηχανισμού διάσωσης, να κριθεί ως παράνομη αντισυνταγματική αυτή η νομική βάση. Εξού και η ανάγκη να τροποποιηθεί η συνθήκη ώστε να αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος ακύρωσης του μηχανισμού από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Όσοι έχουμε πιο φεντεραλιστική άποψη της ε, Ένωσης, ε, θεωρούμε ότι μια τέτοια περιορισμένη μεταρρύθμιση συνθήκης δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, γιατί δεν μας επιτρέπει πιο ε, εις βάθος ολοκλήρωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ενισχύει τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτά τα θέματα. Αυτό βέβαια είναι το ιδεατό. Άλλο όμω το ιδεατό και άλλο το ρεαλιστικό και το εφικτό. Εγώ ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή συντρέχουν οι προϋποθέσεις και είναι πρόσφορο το πολιτικό κλίμα για μια πιο ευρεία μεταρρύθμιση της, συνταγματικής, της ε, συνθήκης. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, ούτως ή άλλως διαπιστώσαμε μια συνταγματική κόπωση. Και συνταγματική κόπωση σημαίνει ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη δεν είναι έτοιμη για ένα νέο άνοιγμα της συνταγματικής διαδικασίας, για μια επανάληψη της συνταγματικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι μια σειρά χωρών με επικεφαλή στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά όχι μόνο, να πούν ναι σε μια συνθήκη, δεν είναι έτοιμες να πούν ναι σε μια συνθήκη που θα ε, δίνει περισσότερε εξουσίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερε δυνατότητε παρέμβαση και περισσότερε εξουσίε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα οικονομικά. Νομίζω ότι είναι μάλλον ψευδέστηση κάτι τέτοιο. Για να μην βαφκαλιζόμαστε ε, λοιπόν με ουτοπίες, θα ήταν αντιπαραγωγικό να προτείνουμε πιο ρηξικέλευτες αλλαγές στη συνθήκη. Κάτι που ε, είναι μάλλον αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Οι πιθανότητες μιας ε, ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης συνθήκη είναι σχεδόν μηδέν, μηδενικές. Και παρά τις φεδεραλιστικές τάσεις που μπορεί να έχουμε ορισμένοι και να είμαστε υπέρ μιας πιο ομοσπονδιακής διακυβέρνησης, θα πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστές και αν δεν αποδειχθεί ότι χρειάζονται και άλλες τροποποιήσεις της συνθήκης, κάτι όμως που προποθέτει συνένεση των κρατών μελών, αν δεν ε, αποδειχθεί αυτή η ανάγκη, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τρέφουμε φρούδες ελπίδες ή ψευδεστήσεις για μια βραχυπρόθεσμη, φιλόδοξη και ευρεία μεταρρύθμιση της συνθήκης. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μορέιρα. Τώρα ζήτησε το λόγο κυρία Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί ο κατάλογος των ομιλητών ε, έχει πολλούς υποψηφίους. Θέλω και εγώ να επανέλθω και να επιμείνω για την ε, ρεαλιστικό χαρακτήρα της απόφασης που έλαβε το Συμβούλιο, το οποίο θεώρησε καθήκον του να ανταποκριθεί σε μια συγκεκριμένη προθεσμία του 2013 και ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή το τέλος του προσωρινού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για ε, τότε. Αντιδρώντας λοιπόν ε, καταρχήν σε αυτή την ε, χρονική προθεσμία και στις νομικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τις αποφάσεις, από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Κάρσρουης, το Συμβούλιο οδηγήθηκε να λάβει μια απόφαση ρεαλιστική. Όπως είπαν και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι, πιστεύω πως δεν θα ήταν πολύ ρεαλιστικό το να προβλέψουμε αλλαγές συνθήκης πολύ ευρύτερες και που θα καταφέρουν ωστόσο να παραμείνουν μέσα σε αυτά τα χρονικά περιθώρια που θα μας επιτρέψουν δηλαδή να ολοκληρώσουμε πριν το 2013. Θα ήταν νομίζω ρεαλιστικό να σκεφτούμε μια αλλαγή συνθήκη που θα περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και χρονικά επίσης περιορισμένο. Το πραγματικό θέμα ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου μας. Γιατί φυσικά πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση της συνθήκης μετά από την ε, θέση εφαρμογή τη συνθήκης ε, Τη Λισαβόνα, Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας παραλληλισμός και αναλογία με άλλες διαδικασίες αναθεώρησης συνθήκες ή άλλους όρους ανάμειξη του Κοινοβουλίου. Ένα Κοινοβούλιο με αρμοδιότητες και με ρόλο πιο ενισχυμένο, χάρη στις συνθήκες της Λισαβόνας, ε, νομίζω θα πρέπει να προβλέψουμε μέσα στη διαδικασία αναθεώρησης που από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει συντόμως όποια και θα είναι το αντικείμενό της. Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα, ότι θα πρέπει να είναι περιορισμένο σε, περιορισμένη σε μια συγκεκριμένο ζήτημα. Θα πρέπει σαφώς να αναμειχθεί το κοινοβούλιο μας, να είναι ένα μάλιστα από τους κύριους πρωταγωνιστές αυτής της αναθεώρησης. Δεν έχω άλλους ομιλητές. Είναι δύσκολο διαπιστώνω να βγάλουμε συμπεράσματα για ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο όντως δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια συζήτηση μια ώρα. Φυσικά θα επανέλθουμε, δεν ξέρω ακριβώς πότε και πού, αλλά σίγουρα το Δεκέμβριο θα υπάρξει νέο συμβούλιο και ο πρόεδρος Μπούζεκ θα συμμετάσχει σε εκείνο το συμβούλιο και άρα ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Μπούζεκ για αυτό το ζήτημα τουλάχιστον ως συντονιστές πριν από το Δεκέμβριο για να εκφράσουμε κάπως πιο συγκεκριμένα όλες τις ανησυχίες και τις προτάσεις μας, όπως αυτές ακούστηκαν απόψε. Ζητώ συγγνώμη που η συζήτηση για αυτό το σημείο έγινε έτσι κάπως απροτήμαστα. Το αίτημα ήταν του συναδέλφου Νταφ να μπει στην ημερήσια διάταξη. Σύμπερ, σας ευχαριστώ. Νομίζω πως συμφωνείτε με αυτό που σας πρότεινα. Και τέλος της συνεδρίασης. Μάλλον να πω πριν να κλείσω ότι ξέχασα στην αρχή, έπρεπε να το κάνω, αλλά κάλλιο αργά παραπότε, να σας θυμίσω πως ε, έχουμε στη γραμματεία μας ένα νέο υπάλληλο. Λέγεται Μέμετς. Δεν είναι παρόν. Α, είναι. Πούντος. Ναι. Α, μάλιστα. Σας χαιρετίζω εξ τη της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή μας ήδη σας γνωρίζει, γιατί νομίζω πως στο παρελθόν έχετε συνεργαστεί με την Επιτροπή τούτη. σα εύχομαι καρποφόρα και αποτελεσματική συνεργασία.